Ladies Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μπορούμε να αρχίσουμε. Θα ήθελα να σας πω εξ αρχής ότι η συνάντηση των συντονιστών θα γίνει στις 11.30 σήμερα. μεταξύ των ομάδων, αν έχω κατανοήσει καλά. Αρχίζουμε λοιπόν εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη σε σχέση με το 3 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την νομική προστασία και κλπ. στην παροχή πρόσβαση από όρους αναβάλλεται και άρα θα στραφούμε στη σύμβαση σχετικά με τις ε, διεθνείς Α, με συγχωρείτε, και το 4, η σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς ασφάλειες επικινητού εξοπλισμού σε σχέση με το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό αναβάλλεται επίσης. Διαφορετικά έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. And we go then και άρα στρεφόμαστε άμεσα στο σημείο υπαριθμών 5 Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών και Διαδικασία Έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής. Η κυρία Γκέριγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να πω ότι οι εργασίες επί του κανονισμού αυτού άρχισαν κατά την προηγούμενη θητεία και τότε ήμουν σε θέση να παρουσιάσω το θέμα, αλλά υπό το νέο κοινοβούλιο, υπό τη νέα θητεία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ορισμένες ιδέες, τους παλαιούς και τους νέους. Σε σχέση με την αλλαγή ως προς τον κανονισμό, ως προς την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Ορισμένες αλλαγές θα επέλθουν στον κανονισμό σε σχέση με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και θα ήθελα να σας πω εγώ, να σας μιλήσω για ορισμένες επιφυλάξεις. Θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή και όσον αφορά ε, την πλειοψηφία των σημείων μπορώ να πω ότι με βρίσκουν σύμφωνοι. Θα ήθελα να σας πω το γενικό πλαίσιο και τις ιδέες μου. Η οικονομική κρίση σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης και του κοινοτικού δικαίου και αυτό σημαίνει υποστήριξη της οικονομίας. Θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να είναι πιο αποτελεσματικό το νομικό σύστημα και ένα από τα μελήματά μας είναι η διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών. Αν δούμε τους υπάρχοντες κανονισμούς, υπάρχουν ορισμένες διαφορές που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά. Μιλώ για μικροδιαφορές και αυτό συνίσταται στη, στο μικρό μέρισμα αυτών των μικροδιαφορών αναχώρες. Βλέπουμε ότι οι αντίδικοι δεν γνωρίζουν πολύ καλά το όλο σύστημα, δεν έχουν δηλαδή πληροφορίες σε σχέση με την επίλυση αυτών των μικροδιαφορών και πολλές φορές ε, πρέπει να επομιστούν έξοδα ταξιδίου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ε, αυτό αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα. Τα επόμενα χρόνια οι μικροδιαφορές θα αυξηθούν και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί, αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των μικροδιαφορών. Άρα, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, ε, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίξαμε το ψήφισμα του Οκτωβρίου του 2011, δηλαδή το ποσοστό προσφυγών για μικροδιαφορές, το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Πολύ λίγοι προσφεύγουν στα δικαστήρια, άρα η διαδικασία θα πρέπει να είναι πιο διαφανής έτσι ώστε να υποβάλλονται προσφυγές, να γίνονται προσφυγές στο δικαστήριο εξάρτητα από το μέρισμα των μικροδιαφορών σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σε σχέση με τις διασυνοριακές μικροδιαφορές θα πρέπει να αυξήσουμε το κατόφλι σε 10.000 ευρώ. Μάλλον το κατόφλι ήταν 10.000 ευρώ, ενώ τώρα θα πρέπει να στραφούμε στη... στο κατόφλι των 2.000 ευρώ. Ίσως το κατόφλι να μην είναι τόσο σημαντικό για τους μικροκαταναλωτές, αλλά τα 2.000 ευρώ είναι ένα ε, καθόλου αμεληταίο ποσοστό. Πρόκειται λοιπόν για ε, ένα κατόφλι που θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Μόνο το 20% των μικροδιαφορών δεν φτάνουν το κατόφλι των 2.000 ευρώ. Αν αυξήσουμε όμως το κατόφλι στα 10.000 ευρώ τότε θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και με αυτές τις διασυνοριακές μικροδιαφορές. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το κατόφλι έτσι ώστε να αυξήσουμε και τον αριθμό των ΜΜΕ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό, αυτό το νέο δηλαδή ε, νομικό μέσο. Και βεβαίως... Και φυσικά θα γίνουν και αποταμιεύσεις και εξοικονομήσεις. Βεβαίως θα επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των, ε, της αντιμετώπισης των μικροδιαφορών. Όμως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πολύ περισσότεροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικά μέσα αποστολής πληροφοριών και τεκμηρίωσης. Αυτή τη στιγμή η επικοινωνία μεταξύ των ε, ε, διαδίκων και των ε, δικαστηρίων δεν είναι επαρκής, ιδιαίτερα διασυνοριακά και όταν μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στο μέλλον, εάν δεν, μάλλον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αυτό αποθάρρυνε τους διαδίκους από τη χρήση αυτής της διαδικασίας. Θα πρέπει να μπορούμε να αποστέλουμε πληροφορίες και να λαμβάνουμε πληροφορίες και ηλεκτρονικά. Γι' αυτό η Επιτροπή και η Επιτροπή μπορεί να λάβει ή να στείλει ε, τεκμηρίωση. έτσι ώστε να υπάρχει και η κατάλληλη εποπτεία της διαδικασίας. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να συσταθεί ένα σύστημα πληροφόρησης των διαδίκων για να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσφυγή τους, δηλαδή ένα σύστημα ε, ιχνηλάτησης. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο της ε, τηλεδιάσκεψης. Αν δείτε τις διαδικασίες αυτές μικροδιαφορών, η γραπτή διαδικασία ε, είναι σχεδόν αποκλειστική. Δεν υπάρχει επακροατηρίου διαδικασία. Όταν υπάρχει θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το μέσο της τηλεδιάσκεψης, διότι νομίζω ότι θα ήταν κάτι το πολύ θετικό, γιατί ακριβώς εξοικονομείται χρόνος. αλλά ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος ε, για να ε, διατεθεί αυτός ο εξοπλισμός σε ορισμένα δικαστήρια που δεν τον διαθέτουν. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Στη δική μου χώρα, στην Πολωνία, ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους ε, η πλειοψηφία των δικαστηρίων θα διαθέτει αυτό τον τεχνικό εξοπλισμό και φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε ένα όριο για τα δικαστικά έξοδα. Τα δικαστικά ε, έξοδα είναι δυσανάλογα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ε, υψηλά 10% της συνολικής αξίας των μικροδιαφορών και αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγων προσφυγής για μικροδιαφορές, διότι τα δικαστικά έξοδα είναι αρκετά υψηλά. Θα θέλαμε λοιπόν να γίνει διευθέτηση μικροδιαφορών και με άλλους τρόπους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα μέγιστο όριο δικαστικών εξόδων που αρχίζουν από τα 40 ευρώ, γιατί αν είναι πολύ υψηλά θα ε, αποθαρρύνουν τους πολίτες. Γιατί αν τα δικαστικά έξοδα είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τη μικροδιαφορά, οι πολίτες δεν θα προσφύγουν στα δικαστήρια. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει δικαστική εκπροσώπηση. Υπάρχουν ορισμένε εταιρείε και επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό και σε αυτό τον παράγοντα, διότι γνωρίζουν ότι οι πελάτες τους ε, δεν θα προσφύγουν αν πρόκειται για μικροδιαφορά και τα δικαστικά έξοδα είναι πολύ υψηλά. Εάν ε, μιλάμε για μία προσφυγή της τάξης των 200 ευρώ, εάν τα δικαστικά έξοδα είναι υψηλά, τότε ο πολίτης δεν θα προσφύγει. πολύ λαμβάνουν υπόψη αυτό τον παράγοντα των υψηλών δικαστικών εξόδων. Μία άλλη πρόταση της Κομισιόν είναι να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν κάποιο σύστημα που επιτρέπει στους πολίτες να καταβάλουν τα ε, δικαστικά έξοδα εξ αποστάσεως. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, διαφορετικούς τρόπους πληρωμής δικαστικών εξόδων. Και αν ο μόνος αποδεκτός τρόπος είναι τα εμβάσματα ή τα μετρητά, τότε τα δικαστικά έξοδα, εάν είναι υψηλά, ε, τότε ο ενάγων θα πρέπει να προσλάβει δικηγόρο γι' αυτό. Εάν λοιπόν μπορούν να καταβληθούν τα δικαστικά έξοδα εξ αποστάσεως, αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο τεχνικής υφής ζήτημα αφορά το, τα έξοδα μετάφρασης. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει υποβληθεί σε σχέση με την νομοθεσία, αλλά πολλές φορές υπάρχουν πολύ ε, δύσκολες φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν και μόνο ένα μέρος ε, της φόρμας είναι σημαντικό, που αφορά τη, το διατάφτα και γι' αυτό θα πρέπει μόνο αυτό το τμήμα της απόφασης να μεταφραστεί και όχι ολόκληρο το έγγραφο της απόφασης, διότι αφορά πολύ υψηλά έξοδα. Πρόκειται για το 4-3 που αφορά την ουσία της απόφασης, το διατάφτα που είναι και το μόνο που θα πρέπει να μεταφραστεί. Επίσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα, πώς θα πρέπει να καταβληθούν και επίσης πληροφορίες συμπλήρωσης της φόρμας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαθέτουμε αυτές τις πληροφορίες για την διαδικασία μικροδιαφορών και επίσης η, συμπλήρωση της φόρμας είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ε, στοιχεία. Υπάρχουν δύο τύποι εναγόντων, τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις. Υπάρχει το όριο, το κατόφλι των 2.000 ευρώ για τις ε, αγωγές, αυτό αρκεί για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά όταν μιλάμε για αύξηση κατοφλίου στις 10.000, αυτό μπορεί να ευνοήσει τις επιχειρήσεις. Άρα οι μικρομεσές θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολύ χρήσιμο μέσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, madam. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο να πάρει το λόγο για να σχολιάσει. The commission, yes. Η Commission. Oh, yeah, Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα την παρουσίαση και διάβασα το έγγραφο με μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαι νέος Ευρωβουλευτής. Ανακαλύπτω σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, αυτή τη διαδικασία κι εγώ. Νομίζω ότι οι προτάσεις που ζητάμε, που κάνουμε μάλλον, πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση και δεν φύγουν το, την ουσία, τον πυρήνα της εθνικής νομοθεσίας, αλλά διευκολύνουν την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών που είναι όλο και περισσότερες. Και αυτό προς το συμφέρον των πολιτών. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Κάποια νούμερα αναφέρονται στην έκθεση. Λέμε π.χ. ότι στην Ισπανία είχαμε χίλια αιτήματα ε, το 2012 για αυτή τη διαδικασία και μόνο τρία στη Βουλγαρία. Τα νούμερα αυτά μας φαίνονται πολύ λίγα. Λάθος κάνω. Ή αυτή η διαδικασία η οποία φαίνεται τόσο ενδιαφέρουσα ε, χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο μέχρι τούδε. Και αν ναι, τι προτείνετε; πολύ συγκεκριμένα, ούτω ώστε να γίνει πιο πλατιά γνωστή και να χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Does the Commission wish to, to comment? Η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you uh, for giving me. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο να απαντήσω στις ερωτήσεις. Για αυτό το θέμα του αριθμού, το, του μικρού αριθμού των ετοιμάτων για τη χρήση αυτής της διαδικασίας. Εμείς το έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα αρκετά νωρί. Το καταλάβουμε ότι υπάρχει και λάβουμε κάποια μη νομοθετικά μέτρα, ούτω ώστε να αυξήσουμε την δημοτικότητα εντό αγωγικών του μέτρου αυτού, τη διαδικασία αυτή. Ετοιμάσαμε συγκεκριμένους οδηγού προ του επαγγελματίε και άλλου οδηγού για του καταναλωτέ, ούτω ώστε να μάθουν πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία μέσω αυτών των εγχειριδίων. Είδαμε ότι η διαδικασία χρησιμοποιείται λίγο, σχετικά θα έλεγα, και λόγω κάποιων νομοθετικών εμποδίων που υπάρχουν. Αυτό βρήκαμε, σε αυτό καταλήξαμε. Τα στοιχεία της πρότασης που ανέφερε η συγγήτρια συνιστούν και εμπόδιο Παραδείγματος χάρη το χαμηλό κατώτατο όριο. Περιορισμένος ορισμός των διασυνοριακών υποθέσεων. Δηλαδή, περιορίζει ο ορισμός ήδη. Και έλλειψη ενημέρωσης και βοήθειας προς τους διαδίκους, προς τα μέρη. Πέρα από αυτά που ανέφερα ως παραδείγματα μη νομοθετικών μέτρων, επίσης, Ήρθαμε σε επαφή με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, που δίδουν συμβουλέ για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικρών Απαιτήσεων. Και τώρα έχουμε λάβει και επιχορηγήσεις για αυτή την δραστηριότητα, δηλαδή να δώσουμε ενημέρωση στους καταναλωτές για τις δυνατότητε και τους τρόπους χρήσης αυτής της διαδικασίας μικρών πληρωμών. Ε, e, Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι έρευνες που έκανε η Κομισιόν δεν είναι πλήρης. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου τα άτομα που έχουν πέσει θύμα Απλώς δεν μιλάνε για το πρόβλημα. Και επομένως τις περιπτώσεις αυτές δεν τις καταγράφουν οι στατιστικές. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στη συζήτηση που έγινε στο φόρουμ στο ίντερνετ. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια επιχείρηση Χ, η οποία δεν υπάρχει γιατί έκανε πολυάριθμες α, προσπάθειες α, κατάχρησης, ας πούμε, ε, μετά εξαφανίζεται και χρησιμοποιεί άλλο όνομα για να πουλήσει τα εμπορεύματά της. Όταν μιλάμε για την ψηφιακή αγορά, όταν μιλάμε για την ανάγκη υποστήριξης της οικονομίας μας, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί πιο ευρέως, βλέπουμε ότι όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα διαδικασία, που ο βασικός της στόχος είναι να περιοριστούν οι καταχρήσεις και οι παραβιάσεις, ε, είναι απαραίτητο να γίνει πραγματική χρήση Αυτέ οι διαδικασίε, αντίστοιχε μάλλον διαδικασίε, υπάρχουν σε πολυάριθμε χώρε, αλλά όχι εναρμονισμένε. Έτσι. Αυτή όμω είναι υπέρτατη ανάγκη στην ενιαία αγορά. Να υπάρξει εναρμόνιση αυτή τη διαδικασία και να εισαχθεί η διαδικασία όταν δεν υπάρχει, σε χώρε που δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ πρακτική λύση που θα εξυπηρετήσει του πολίτε. Θα έχουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια χάρη σε αυτή τη διαδικασία και θα αισθάνονται ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαία αυτή η αναδιατύπωση και εμείς θέλουμε η δικαιοσύνη να είναι πολύ κοντά στον πολίτη. Αυτή η διαδικασία σίγουρα είναι ευεργετική. Πέραν όμως από όλες τις επιφυλάξεις που θα μπορούσαμε να έχουμε και σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνολική αξία αυτής της ε, διαδικασίας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολλά φυσικά πρόσωπα τα οποία ε, εργάζονται σε διάφορες ε, χώρες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαδικασία επίλυσης ε, μικροδιαφορών. Γι' αυτό θα ήθελα να μην ισχύει αυτό το κατόφλι μόνο για ΜΜΕ. Στη Ρουμανία έχουμε αυτή την απλουστευμένη διαδικασία που αφορά την γραπτή φάση και μπορεί να υπάρξει και μία διαδικασία επακροατηρίου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το κατόφλι θα μπορούσε να είναι υψηλότερο και για τις ΜΜΕ ε και όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Ίσως θα μπορούσαμε να ταχθούμε και στα 15.000 ευρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούντα για τα σχόλιά σας. Πρέπει να πω ότι και εγώ σκέφτηκα την αύξηση του κατοφλίου. Είχα αυτή την πρόθεση. Πέραν των 10.000 ευρώ δηλαδή. Αλλά θα δούμε πώς θα αντιδράσει και το Συμβούλιο σε πρώτη φάση στα 10.000 ευρώ. Από κάποιες ε, ανεπίσημες συζητήσεις που είχαμε μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τα 10.000 ευρώ ως ε, κατόφλι. Νομίζω ότι είναι για μένα τουλάχιστον τα 10.000 ευρώ είναι το ελάχιστο όριο ώστε να μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να προσφεύγουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αλλά ε, σε κάθε περίπτωση αν μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτήν τη θέση θα μας βοηθήσει τη διαπραγματεύση μας με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Διότι ε, θέλουμε προφανώς το έγγραφο αυτό να υποβληθεί σε επεξεργασία το συντομότερο δυνατό. Ε, ενδεχομένως και επί Ιταλικής Προεδρίας ακόμη. Ή τουλάχιστον να έχουμε μια διεξοδική ανάλυση Τη κατάσταση. Αυτή που η παρουσίαση που έκανα σήμερα είναι μια πρώτη παρουσίαση ε, της εισηγησής μου, της ε, έκθεσής μου και βεβαίως ε, θα μπορείτε να υποβάλλετε και τροπολογίες στη συνέχεια να ψηφιστεί στην Επιτροπή η συμβαστική αυτή εκδοχή του κειμένου και στη συνέχεια θα πάμε σε διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε εντός του, του έτους, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο μία διαδικασία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Ε, όπως είπα για τα δικαστικά έξοδα πρέπει να υπάρχει ε, κάποιο ανώτατο όριο διότι αυτό που θέλουμε είναι να μην αποθαρρύνονται οι πολίτες από το να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος κύριε Κομοντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πρακτική εμπειρία στο παρελθόν, νομίζω ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διασυνοριακές ε, διαφορές. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Το άρθρο 18 ε, της αναθεώρησης ε, της διαδικασίας ορίζει ότι τα κράτη-μέλη θα δώσουν στοιχεία για την αναθεώρηση. Πολλές φορές η αναθεώρηση αυτή διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή αν υπάρχουν πληροφορίες για τη διαδικασία που ακολουθείται, που ισχύει ήδη στα κράτη-μέλη. Διότι ε, ενδεχομένως θα πρέπει και αυτό το ζήτημα να το λάβουμε υπόψη μας στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Can the commission react? Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ερώτηση. Δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια της ε, διαδικασίας αναθεώρησης, που είναι μια πολύ ειδική διαδικασία. Δεν πρόκειται για κάποια εθνική ε, προσφυγή. Αφορά μόνο τον, ε, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ο διάδικος μπορεί να ζητήσει αναθεώρηση. Δυστυχώς τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτής της διαδικασίας στα κράτη-μέλη δεν είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρουμε σε πόσες περιπτώσεις δηλαδή οι εναγόμενοι ζητούν αυτή την ειδική διαδικασία και πόσο τελικά διήρκησε ε, για πόσος χρόνος χρειάστηκε για την έκδοση απόφασης. Η αλλαγή στο άρθρο 18 που προτείνουμε είναι τεχνικής φύσης και αποσκοπεί στο να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση που χρησιμοποιείται στη διάταξη με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται ήδη τη νέα διατύπωση που χρησιμοποιείται ήδη σε άλλους κανονισμούς. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ευθυγραμμίσουμε βεβαίως και κατά περίπτωση τις διατάξεις ε, όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ε, αστικές διαφορές. Και αυτή η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών πρέπει να είναι μια ταχεία διαδικασία. Είναι ήδη επιταχυμένη, αλλά θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι ιδιαίτερα αυτή αυτή αυτό το στοιχείο εφαρμόζεται με έναν αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Κανονικά θα περνούσαμε τώρα στο σημείο 6, αλλά επειδή πρόκειται για σημείο που θα γίνει ψηφοφορία και επειδή συνήθως οι ψηφοφορίες στην Επιτροπή μας γίνονται γύρω στις 10 και επειδή ο κύριος Ντούντα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ο εισηγητής δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, θα πρότεινα να παρακάμψουμε το συγκεκριμένο σημείο και να περιμένουμε μέχρι τις 10, οπότε και θα έρθει ο κύριος Ντούντα. Ε, Για το 7 δεν είναι εδώ δυστυχώς μαζί μας ακόμη ο γραμματέας του δικαστηρίου, οπότε θα πρότεινα να παρακάμψουμε και αυτό το σημείο και να πάμε στο σημείο 8 όπου είναι μαζί μας η εισηγήτρια η κυρία Ντελβό οπότε ε, έχει το λόγο η κυρία Ντελβό Ευχαριστώ Πρόεδρε Και εγώ είμαι νέα ε, βουλευτής και αυτό το θέμα της απλούστευσης ε, των δημοσίων εγγράφων έχει ένα ιστορικό. ανέλαβα το θέμα από τον κύριο Ραπκάη που δεν είναι πια ευρωβουλευτής. Γιατί πρόκειται για τα νέα μέλη. Υπάρχουν όλο ένα και περισσότεροι πολίτες που ζουν σε κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος μέλος προέλευσης και θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα των πολιτών ανά την Ευρώπη και πολλές φορές όταν μεταβαίνετε από το ένα κράτος σε ένα άλλο θα πρέπει να τηρήσετε μία διαδικασία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013 πρότεινε ένα κανονισμό και το Κοινοβούλιο ε, προέβη σε μια πρώτη ανάγνωση το Δεκέμβριο του 2013. Μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση ε, της Επιτροπής έχει ως εξής. Την διαγραφή ε, μετά της διαδικασίας μετάφρασης. Ε, ως προς τις ληξιαρχικές πράξεις, ε, θανάτου, συμβίωσης, γάμου, γέννησης, μπορούμε να πούμε ότι δεν αφορά ε, μόνο τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τις επιχειρήσεις. Άρα, πολλές φορές δεν χρειάζεται ε, μετάφραση, ιδιαίτερα όταν κανείς μεταβαίνει σε ένα άλλο κράτος μέλος. Σε σχέση με την πιστοποίηση εγγράφων, η πρόταση ε, αφορά την απαλυφή αυτής της υποχρέωσης. Αν δηλαδή υποβάλετε τα ε, πρωτότυπα έγγραφα, δεν χρειάζεται να υποβάλλεται ε, ένα πιστοποιητικό θεωρημένο. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτή η πιστοποίηση που είναι ε, δαπανηρή. Το ίδιο αφορά και τις ε, μεταφράσεις. Όσον αφορά τις μεταφράσεις, πολλοί ζητούν ε, θεωρημένες μεταφράσεις και πολλές φορές ε, η πιστοποίηση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από ορισμένα κράτη-μέλη. Άρα δεν χρειάζεται ε, μετάφραση πιστοποιημένη, απλώς μία μετάφραση. Και αν η χώρα υποδοχής έχει αμφιβολίες ε, σε σχέση με τη μετάφραση, τότε μπορεί να ζητήσει θεωρημένη μετάφραση. Το τρίτο θέμα είναι ο φόβος της απάτης, δηλαδή αν υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μέλων μέσω της διαδικασίας εσωτερικής αγοράς ΙΜΗ είναι το ακρόνιμο και αυτό αφορά και τα προσόντα και τα διπλώματα. Και επίσης θα πρέπει να οριστεί ένα πολύγλωσσο έγγραφο, δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ζητήσει να του δοθεί ένα πολύγλωσσο πιστοποιητικό που θα έχει την ίδια αξία με το εθνικό. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι προτάσεις αφορούν την πιστοποίηση εγγράφων. Δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζονται αυτόματα, απλώς υποβάλλονται στη χώρα υποδοχής. Στη συνέχεια το κράτος μέλος, το νέο κράτος μέλος μπορεί να αναγνωρίσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξήσει τον αριθμό των δημοσίων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πέρα από τις ληξιαρχικές πράξεις ή τις πράξεις ε, οικογενειακής κατάστασης έχει ε, λάβει υπόψη και έχει επεκτείνει και στα πιστοποιητικά ε, δε, της ε, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πράξεις και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες ως προς το αυθεντικό χαρακτήρα του εγγράφου μπορεί να ζητήσει θεωρημένη μετάφραση, αλλά σε αυτή την περίπτωση το κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να αναλάβει και τα έξοδα. Αυτά επί του κανονισμού. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε εάν γίνουν αλλαγές ε, στο έγγραφο σε σχέση με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία τότε θα αναπαιμφθεί αυτό το έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών προχωρούν. Η Ιταλική Προεδρία ανακοίνωσε ότι θέλει να προχωρήσει στα θέματα αυτά και αναμένουμε μια νέα πρόταση τον Δεκέμβριο. Βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη ίσως ε, περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει παραχάραξη μητρών και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη αν θα υπάρξει αυτή η προέκταση ή επέκταση. Περιμένουμε την, ε, αναμένουμε την πρόταση του Συμβουλίου Υπουργών και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση τη στιγμή που θα έχουμε και την τελική θέση του Συμβουλίου και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τη δεχτούμε και κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Έτσι κι αλλιώς διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν. Περί αυτού πρόκειται και θα ήθελα τέλος να αναφέρω το εξής. Εγώ τώρα ανακαλύπτω αυτό τον κανονισμό και θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ καλό βήμα προς τα μπρος για τους πολίτες. Τουλάχιστον τους πολίτες που μεταβαίνουν από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο μπορούν να ευεργετηθούν από αυτόν τον κανονισμό, διότι πρόκειται για πραγματική απλούστευση για την αναγνώριση των δημοσίων εγγράφων και αυτό αφορά και τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ε, εργαστούν ε, διασυνοριακά. Άρα μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία διασυνοριακής συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού ζητήσω τα σχόλιά σας, να σας ζητήσω αν θα μπορούσαμε να ανακοινώσουμε ήδη τα ονόματα των όσων συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Ε, δεν ξέρω, λέει η κυρία Ντελβό, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Οπότε δεν, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει κάτι. Φυσικά, ναι, καλό θα ήταν να ξέρουμε ποιο θα είναι ε, στην, ε, σε αυτή την ομάδα διαπραγμάτευσης, αυτή την αντιπροσωπεία, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ωραία, τότε θα το συζητήσουμε αργότερα. Ο κύριος Ράντεβ ζήτησε το λόγο. Благодаря, господин председател. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι η απλοποίηση αυτών των διοικητικών τυπικών διδικασικών για να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κληροφορίας των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, το δικαίωμα εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις, η ελευθερία ε, παροχής υπηρεσιών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες και στην απουσία διμερών ε, ε, συμφωνιών Πολλέ φορέ οι διαδικασίε αυτέ είναι πάρα πολύ χρονοβόρε και δύσκολε. Οπότε οι διαδικασίε θα απλουστευτούν σίγουρα για πάρα πολλού ε, πολίτε. Είμαι πολύ χαρούμενο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για αυτό το ζήτημα. Ε, ελπίζω να ε, ευοδοθούν και οι διαπραγματεύσεις ε, με, τους, με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ως δικηγόρος πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της νομικής ασφάλειας και των και των ωφελών που θα προκύψουν. Ελπίζω ε, μέχρι το τέλος του χρόνου να καταφέρουμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καρίμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για αυτήν την σε βάθος ε, παρουσίαση του θέματος και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να τύχει της υποστήριξης του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η ίδια η πρόταση μάλλον δεν εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Το ζήτημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε επί της αρχής να υπάρχει μεγάλη συμφωνία, θα, επειδή ακριβώς είναι κάτι που θα το χαιρετήσουν οι πολίτες, το ζήτημα που μας απασχολεί εδώ είναι το πεδίο ισχύω. Ε, γιατί όταν αρχίσαμε να ε, ασχολούμαστε με έγγραφα που δεν είναι απαραίτητος ε, επίσημα έγγραφα, για παράδειγμα έγγραφα που εκδίδει κάποιο πανεπιστήμιο, τότε αρχίζουμε να διευρύνουμε τόσο πολύ το πεδίο που τελικά θα αυξηθεί και το άχθος. Από τις ε, εργασίες που είχαμε κάνει με τον προηγούμενο εισηγητή φάνηκε ότι τελικά υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη που ε, αποδέχονται ε, τέτοιου είδους έγγραφα και που ξεκινούν τις έρευνες μόνο αν υπάρχουν υποψίες ή αν υπάρχουν υποδείξεις ότι το έγγραφο που έχει υποβληθεί δεν είναι αυθεντικό. Αν υπάρξει μια τέτοια συζήτηση στις διαπραγματεύσει. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να, να τύχουμε υποστήριξη όσον αφορά την εντολή Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Θα συνεχίσουν οι διαδικασίες και θα χρησιμοποιήσουμε τους κλασικούς διοικητικούς μηχανισμούς. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν ε, γίνει σημαντικά βήματα, θεωρώ και εγώ, για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και τα συμφέροντά τους. Παράλληλα, από την εμπειρία μου ως δικηγόρος, μου προκύπτει μία απροθυμία να δεχτώ το πεδίο εφαρμογή της διαδικασίας. Μην ξεχνάμε το δίκτυο ασφαλείας που θα πρέπει να έχει αυτό το αστικό δίκτυο. Και βεβαίω θα πρέπει το δίκτυο αυτό να απλώνεται και στους συμμετέχοντες σε αυτό το δίκτυο. μιλήσαμε για τι άδειε οδήγηση, ο εισηγητή δηλαδή. δεν έχω, δεν μ' αρέσει αυτό, γιατί οι προποθέσει για να πάρει κανεί άδεια οδήγηση, να βγάλει κανεί άδεια οδήγηση, ε, διαφέρουν από κράτο μέλο σε κράτο μέλο και είναι πολύ εύκολο να έχει κάποιο πλαστά έγγραφα. Πλαστή δηλαδή. Ε, μην ξεχνάμε λοιπόν ποια είναι τα, τα έγγραφα τα οποία θα υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό αυτό το πεδίο, να μπει οποιοδήποτε έγγραφο μέσα θα πρέπει να αποφύγουμε περιπτώσεις όπου στα πλαίσια αυτού του αστικού δικτύου διακυβεύεται η ασφάλεια του πολίτη και τίθεται ένα αμφιβόλο. Θα πρέπει να θέσουμε κάποια ποσά επίσης, να τα προσδιορίσουμε για το κόστος της μετάφρασης. Αυτή είναι μια πιθανή λύση. Δεν θα πρέπει όμως να θυσιάζουμε την ασφάλεια των πολιτών στη διαδικασία αυτή. Thank Ο κύριος Μαρινάου Πίντου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερασπίζομαι, καταρχήν, όλα τα μέτρα που προωθούν και διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Αυτή η Ευρώπη οικοδομήθηκε στα πλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίων, χρήματος κεφαλαίων δηλαδή, και ελεύθερης κυκλοφορίας των επιχειρήσεων. Εγώ, η Ευρώπη που υπερασπίζουμε είναι η Ευρώπη η οποία θα πρέπει να δώσει, να βάλει στην καρδιά της, στο κέντρο της, στον πυρήνα της, τους πολίτες. Μια Ευρώπη η οποία βοηθάει τους πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τώρα έχουμε μετανάστες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μετανάστες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βήμα το θεωρώ ως ένα ακόμα βήμα για την προώθηση μιας ελευθερίας η οποία δεν έχει υλοποιηθεί 100% στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ο σημερινός κόσμος είναι ένας επικίνδυνος κόσμος, γεμάτος προβλήματα και, και κινδύνους. Τα άτομα τα οποία φύγουν την ασφάλεια της, ε, την ασφάλεια της Ευρώπης ε, συχνά χρησιμοποιούν έγγραφα τα οποία δεν προκαλούν καμία υποψία στις ευρωπαϊκές αρχές. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεν προκαλούν ποτέ αυτά τα άτομα ε, και τα έγγραφά τους, ας πούμε, ε, καμία υποψία. Είναι τέλεια. Μοιάζουν με τα γνήσια. Θα πρέπει, λοιπόν, αυτό το μέτρο να πάει λίγο παραπάνω. Έχουμε, μιλάμε για την Ευρώπη των ε, Γερμανών, των ε, Ιταλών, των Ισπανών, των Ελλήνων κτλ. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα με την ίδια ελευθερία, με τις ίδιες αρχές. Και να σεβόμαστε αυτή την αρχή της ελεύθερη κυκλοφορίας κεφαλαίων αγαθών και προσώπων με τον ίδιο τρόπο. Είναι η ίδια ελευθερία. Η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την κυρία Ντελβό, η οποία ε, Μα έδωσε μια ενδελεχέστατη εξήγηση για το στόχο που θέλουμε να υλοποιήσουμε και το που έχει φτάσει το πράγμα. Να σα ενημερώσω για το πώ προχωρούν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Καταρχά να σα πω ότι η Κομισιόν καλωσορίζει θερμά, καλωσορίζει μάλλον και χαίρεται για αυτή την υποστήριξη ε, που είχε εκφράσει και το παλιό Ευρωκοινοβούλιο αλλά και το σημερινό. Είναι σημαντική πρόταση για τους πολίτες, είναι σημαντική πρόταση και για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται και αυτές από αυτές τις διατυπώσεις. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ κυρίως τους πολίτες έχουμε στο μυαλό μας, γι' αυτό χρησιμοποίησαμε και αυτή τη νομική βάση. Μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή για των πολιτών. Αυτή είναι στην, στη βάση αυτής της ε, πρότασης και χαιρόμαστε που μας υποστηρίζετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι Υπάρχει ένα κοινό όραμα, να το πω έτσι, Ω προς το στόχο που επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε με αυτή την πρόταση. Τούτου λεχθέντος. Υπάρχουν κάποια καθόδη σημεία όπου προσκρούει η συζήτηση και δεν τα έχουμε επιλύσει. Η Ιταλική Προεδρία όμως επιθυμεί να προωθήσει το φάκελο αυτό, τις συζητήσεις αυτές και σκοπεύει να υπάρχει η γενική προσέγγιση έτοιμη το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Συγγνώμη, ε, δικαιοσύνης, και εσωτερικών υποθέσεων. Επίση, θα γίνει μια συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο, τόσο ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα. Ε, αυτό σκοπεύει να κάνει η Ιταλική Προεδρία. Τώρα, να σα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τι δυσκολίε. Το πρώτο θέμα είναι το πεδίο εφαρμογή που απασχολεί. Αν θα θυμάστε, η πρόταση τη Κομισιόν κάλυπτε βασικά στοιχεία δημοσίων εγγράφων για τους πολίτες και κάποιους τομείς που επηρεάζουν την ε, ζωή των επιχειρήσεων. Ε, κτηματομεσίτες, ε, πνευματικά δικαιώματα και κάποια έγγραφα στα πλαίσια του εταιρικού δικαίου. Από τις συζητήσεις που προκύπτουν στο Συμβούλιο είναι σαφές ότι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου εστιάζεται πολύ περισσότερο στα αστικά έγγραφα, αποκλειστικά. Ένα άλλο στοιχείο της ε, πρώτης Κομισιόν ήταν ε, η εισαγωγή αυτών των πολύγλωσσων τυποποιημένων εγγράφων. Αυτό μάλιστα το επικύρωσε και η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Αυτά τα έντυπα, τα πολύγλωσσα, θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ανεξάρτητα. Ε, παράλληλα προς τα πρωτότυπα. Το καλό είναι ότι γλιτώνουμε έξοδα μετάφρασης. Όλοι κάποιοι πολίτε που βρίσκονται σε τέτοια διασυνοριακή εντό εγωγικών κατάσταση, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσαν να ζητήσουν αυτό το έντυπο, το πολύγλωσσο, αν ξέρουν ότι στο μέλλον, α πούμε, θα μεταβούν σε ένα άλλο κράτο μέλο. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο τη πρόταση τη Κομισιόν και το δέχτηκε σε μεγάλο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το υποστήριξε ε, πολύ περισσότερο γιατί ο αριθμός των ε, τέτοιων πολύγλωσσων τυποποιημένων εγγράφων που προσαρτούνται στην πρόταση αυξήθηκε με την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο ήθελε περισσότερα λέει, τέτοια έγγραφα. Στο Συμβούλιο όμως το βλέπει πιο περιοριστικά το πράγμα, ε, το πράγμα αυτό. Η συζήτηση είναι δύσκολη για αυτό το σημείο. Και κάποια κράτη-μέλη έχουν τη θέση ότι δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ανεξάρτητα αυτά τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα από τα πρωτότυπα. Αλλά θα πρέπει να προσαρτώνται στα πρωτότυπα ε, έγγραφα. Κάτι που αλλάζει κατά τη την πρόταση της Κομισιόν. για τις α, γνήσιες μεταφράσεις, για τις βεβαιωμένες γνήσιες μεταφράσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να τις ζητάνε αυτές τις μεταφράσεις των εγγράφων πολύ πιο εύκολα και να μην βασίζονται στην ε, μετάφραση των, εγγράφων που, που άρα έχουν οι πολίτες. Και ένα άλλο τεχνικό θέμα, αλλά σημαντικό για τα κράτη-μέλη, είναι η σχέση μεταξύ της πρότασης της και διαφόρων διεθνών συμβάσεων όπως η σύμβαση ΣΥΕΚ, η συμβάση ΣΥΕΚΑ. Τέλος. Για να σταματήσω κιόλα. Τα εργαλεία πληροφορικής που συνοδεύουν και εξασφαλίζουν τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αν θυμάται στην πρόταση, η πρόταση προέβλεπε ότι θα υπάρχει ένα μηχανοκρατωμένο εργαλείο, το ΙΜΗ, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη και τις αρχές τους να επικοινωνούν εύκολα σε περίπτωση ερωτήσεων για κάποια συγκεκριμένα έγγραφα ή απορριών. Διάφορα κράτη-μέλη θα ήθελαν να περάσουμε σε μια επόμενη γενιά ε, λύσεων πληροφορική και επομένως γίνεται μια αρκετά τεχνική συζήτηση γύρω από το σημείο στο Συμβούλιο. Τέλο πάντων, εμεί είμαστε επεπισμένοι ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδο αυτό και σα βεβαιώνω ότι η Κομισιόν είναι πανέτοιμη για να υποστηρίξει όσο μπορεί την προσπάθεια, ούτω ώστε η αρχική φιλοδοξία τη πρόταση και η σαφή θέση του Κοινοβουλίου, όπω προέκυψε από την πρώτη ανάγνωση, να διατηρηθούν. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαδικασία είναι πολύ ικανοποιητική. Θα ενισχύσουμε έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρώπη και οι πολίτες θα δεχτούν πιο εύκολα την Ευρώπη έτσι. Θα, μειώσουμε τις ε, γραφειοκρατικές ε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Μία ερώτηση θα θέλω να κάνω τώρα. Αν όλα αυτά τεθούν σε ισχύ, προβλέπουμε να γίνει μια αξιολόγηση του κανονισμού. Προβλέπετε κάτι τέτοιο. Υπάρχει... Υπάρχουν και όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των εγγράφων. Δεν θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Η Κομισιόν θα ήθελε να αντιδράσει. Ευχαριστώ. είναι σαφές και είναι καλή η πρακτική το να γίνεται μια αναθεώρηση των ε, νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εδώ. Προβλέπεται μια τέτοια αναθεώρηση. Φυσικά η ακριβής ε, διατύπωση μπορεί να συζητηθεί για να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα θέματα πιο πολύ αν θέλετε. Αλλά εμείς είμαστε απόλυτα ανοιχτοί να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία αναθεώρησης η οποία θα λειτουργήσει ομαλά. Ευχαριστώ και εγώ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Ντελβό, να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση νομίζω και βλέπω ότι το νέο κοινοβούλιο έχει την ίδια προσέγγιση με το παλιό κοινοβούλιο. Είμαστε υπέρ λοιπόν αυτού του σχεδίου για να διευκολύνουμε ακριβώς την ελεύθερη κυκλοφορία Επίσης, καταλαβαίνω απόλυτα το φόβο που έχουν κάποια κράτη-μέλη για ένα, από ένα υπερβολικά διευρυμένο πεδίο εφαρμογή. Μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με αυτά τα κράτη-μέλη για το πεδίο εφαρμογή και σε αυτήν την περίπτωση η ρήτρα αναθεώρηση θα μας επιτρέψει, νομίζω, να προχωρήσουμε χωρίς προβλήματα. Η ρήτρα αυτή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αφορά όχι μόνο το πεδίο εφαρμογή και την ασφάλεια, αλλά και τα μέσα τα οποία, και τα εργαλεία τα οποία δημιουργούνται για να καταπολεμηθεί απάτη. Το εργαλείο που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο, είναι ικανοποιητικό ή μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις. Από την άλλη, να σας πω και κάτι άλλο. Να μην υπερβάλλουμε και υπερβολικά ε, για τη σημασία των ε, απατών, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να είναι άμυρο απατών, ε. πάντα υπάρχουν. Πιο αποτελεσματικοί θα ήμασταν αν είχαμε μια συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, νομίζω. Σε ό,τι αφορά τις μεταφράσεις. Το να ζητάμε να πληρώνονται μεταφράσεις. Νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξουμε προσεκτικά. Να κοιτάξουμε προσεκτικά και τη φύση των εγγράφων. Γιατί μεταξύ των εγγράφων που προτείνονται υπάρχουν πολύ απλά έγγραφα. Παραδείγματο χάρη πράξη γέννηση, που μιλάει για την, τον τόπο και τη μερομηνία γέννηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ζητήσουμε μια πιστοποιημένη μετάφραση, επίσημη μετάφραση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση διαβαθμισμένη ανάλογα με την περιπλοκότητα του εγγράφου. Αυτά, Πρόεδρε. Αυτά ένα αναμονή των εξελίξεων για το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε τώρα στο σημείο 6. Ο κύριος Ντούντα επέστρεψε. Οπότε πάμε στο σημείο 6. Αναδιατύπωση του κώδικα θεωρήσεων της Ένωσης. Κύριε Ντούντα, έχετε το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη που άργησα. Πρόκειται για την αναδιατύπωση του κειμένου, οπότε μπορούμε, αφού είναι τεχνικό το ζήτημα, να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Hey, ε, Ωραία. μπορούμε να ψηφίσουμε με ανάταση της χειρός ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μηχανηματάκια μας. Θα πρότεινα να γίνει ε, διανατάσταση της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχή. Κανείς. Οπότε υπερψηφίστηκε. Ε, να προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο 7. Ο λόγος του κύριο Μαρίνια Επίντο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε να κάνουμε με μία πρόταση αναδιατύπωσης ε, καθαρά σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των ε, δικαστών από 28 σε 40. Όπως ξέρετε, πρόκειται, υπάρχει το Γενικό Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Το ίδιο το Γενικό Δικαστήριο ζήτησε την αύξηση αυτή και θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, δηλαδή τροποποιούμε το καθεστώς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνουμε τον αριθμό των δικαστών από 28 σε 40. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια γενική συμφωνία, διαφωνία υπάρχει μόνο ο τρόπος διορισμού αυτών των 12 δικαστών. Οι 28 αρχικοί δικαστές ε, ορίστηκαν ως, ως εξής ε, ένας ανακράτος. Τώρα μιλάμε για επιπροσθέτως 12. Ε, ε, δεν μπορούν να οριστούν από κάθε κράτος γιατί είναι 12 και τα κράτη-μέλη είναι 28. Άρα θα πρέπει να επιλεγούν με βάση κριτήρια καθαρά αξιοκρατίας αυστηρά κριτήρια αξιοκρατίας. Πολλές φορές όμως ε, μιλώντας για αξιοκρατία δεν είμαστε απόλυτα σαφείς. Αυτό που έχει σημασία είναι οι μηχανισμοί που διέπουν τις επιλογές. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να λάβετε υπόψη. Θα έχουμε να κάνουμε με μία δαπάνη 12 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί κάθε δικαστής στοιχίζει ένα εκατομμύριο ετησίως στο γενικό προϋπολογισμό. Επίσης, το επιχείρημα αύξηση από 28 σε 40 είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει να αντιμετωπίσει 1.325 υποθέσεις που εκκρεμούν ήδη από το 2013. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, το 2009 είχαν ε, να αντιμετωπιστούν γύρω στις 1500 υποθέσεις και απέμειναν 193 υποθέσεις που εκκρεμούσαν. Δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το 2010 από τις 693 υποθέσεις εκδικάστηκαν 527, ε, δηλαδή απέμειναν εκρεμείς 211. Το 2011 είχαμε 725 υποθέσεις, ε, δικάστηκαν 714 και είχαμε αρκετές υπολοιπόμενες. Το 2013 εκρεμούσαν 1237. Αυτό σημαίνει ότι το 12 ο μέσος όρος αποφάσεων για κάθε δικαστή ήταν 24. Δηλαδή κάθε δικαστής εκδίκασε 24 υποθέσεις. Το 2013 περάσαμε σε 25 υποθέσεις ανά δικαστή. αν αυξηθούν σε 40 θα μειωθεί ο αριθμός εκκρεμοδικιών και αριθμός υποθέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε δικαστή. Νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνουμε μία σωστή λύση, αλλά θα πρέπει να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Και θα πρέπει να επισκεφθούμε και το ίδιο το δικαστήριο επίσκεψη που ήδη έχει δρομολογηθεί έτσι ώστε να δούμε ε, επιτόπου πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τις, δικασ... τις δυσκολίες του και ούτω καθεξής. Για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, γιατί δεν νομίζω ότι ο αριθμός των υποθέσεων ε, αυτού θα οδηγούσε σε αύξηση των δικαστών. Το ανώτατο δικαστήριο, τον είπα, έχει 11 δικαστές. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι η τεχνική υποστήριξη σε κάθε δικαστή. Αλλά θα πρέπει να γίνει μία ειδική ανάλυση και συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Γι' αυτό θα είναι πολύ σκόπιμη η επίσκεψη που προβλέπετε για να συναντήσουμε τους δικαστές και το προσωπικό γενικότερα, έτσι ώστε αυτή η απόφαση να είναι μια δημοκρατική απόφαση ε, όπου δεν διασπαθίζονται δημόσια, δεν διασπαθίζεται δημόσιο χρήμα και μπορούμε να φτάσουμε στους απότερους στόχους. Ο αριθμός εκκρεμοδικιών είναι υψηλός και σίγουρα δεν ευεργετεί ούτε τους πολίτες ούτε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, εάν υπάρχει καθυστέρηση στη δικαιοσύνη, πάβει να είναι δικαιοσύνη. Εάν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη εν ευθέτω χρόνο, τότε δεν τηρούνται οι συνταγματικές προδιαγραφές και δεν βοηθά την κοινωνία έγκαιρα. Πρέπει να προωθήσουμε τα δικαιώματα του πολίτη και από ανθρώπινη πλευρά και λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, συλλογικές ε, οντότητες. Διαφορετικά υπάρχει πρόσκομα στην ε, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Διαφορετικά ακροτηριάζεται ο πολίτης ως προς την διάσταση της ε, υπηκότητάς του, της οντότητάς του. Θα πρέπει λοιπόν να αποφαίνεται η δικαιοσύνη έγκαιρα έτσι ώστε να φτάνει στους βασικούς της στόχους, γιατί γι' αυτό υπάρχει, αυτό είναι ο λόγος ύπαρξής της. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ζβεύκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρίνιο Επίντο για την εξαιρετικά σαφή παρουσίαση της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είχα την ε, ευχαριστη, την ευχαρίστηση να συνεργαστώ με τον προηγούμενο συγητή στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια λογική, ως κοινοβούλιο, σε μια λογική λύση. Τώρα η καυτή πατάτα είναι βέβαια στα χέρια του Συμβουλίου. Έχουμε συμφωνήσει και εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια ότι το κριτήριο ε, των ε, επαγγελματικών προσόντων θα είναι το σημαντικότερο κριτήριο για τον διορισμό των δικαστών. Και ε, υπάρχει και η αρχή ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν δικαστή ως μέλος του δικαστηρίου. Κανένα κράτος μέλος δεν θα έχει επίσης πάνω από δύο δικαστές. Και αυτό είναι σημαντικό διότι όταν θα προσπαθήσουμε να βρούμε δικαστές στη βάση μόνο των επαγγελματικών προσόντων και όχι στην ε, βάση του, του κράτους μέλους και της υπηκότητας, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με κάποιον περιορισμό αριθμητικό. Πρέπει να επιμείνουμε στη θέση μας και να διασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο δεν θα υπονομεύσει την ε, θέση μας. Φυσικά, έχει προγραμματιστεί μια επίσκεψη στο Λουξεμβούργο που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη τόσο για τα παλαιότερα όσο και για τα νεότερα μέλη της Επιτροπής μας και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να γίνει και μια ανταλλαγή απόψεων. Και θα μπορέσουμε να δούμε από πρώτο χέρι ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι δικαστές. Δυστυχώς, το θέμα που ανέφερε ο κύριος Μαρίνιο όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται για να εκδικαστεί κάθε υπόθεση στο δικαστήριο, ο οποίος γίνεται όλο ένα και περισσότερος, όλο ένα και μεγαλύτερος, εν μέρη και λόγω της αύξησης του αριθμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται βέβαια το γεγονός αυτό και στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο πανευρωπαϊκά ή διασυνοριακά υπάρχουν, προκύπτουν δηλαδή και δικαστικά ζητήματα ως συνέπεια. Και οι διαμάχες πολλές φορές δεν καταλήγουν στα εθνικά δικαστήρια. Αυτοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση των υποθέσεων. Κανείς όμως δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη και το κόστος αυτής της αύξησης. Τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς θα διοριστούν δηλαδή οι επιπλέον αυτοί δικαστές προκειμένου να προκειμένου το δικαστήριο να χειρίζεται ε, γρηγορότερα τις υποθέσεις για να διευκολυνθεί και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν και κάποιες αρκετά φιλόδοξες επιδιώξεις, προσδοκίες από την πλευρά των κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία τόσο του δικαστηρίου όσο και της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος του να έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που καλέσατε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συμμετάσχει σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση, που αποτελεί την επανέναξη της ενασχόλησης μας με το φάκελο αυτό, που έχει ξεκινήσει εδώ και μισή χρόνια. Ξέρετε ότι το 2011 το δικαστήριο έκανε μια πρόταση για αύξηση, ας πούμε, των υποθέσεων και με τις εξηγήσει που έδωσε. Μάλιστα ήταν, ε, είχε έρθει εδώ το, το πρόεδρος, ο κ. Κουρίζη, να παρουσιάσει την πρόταση. Είχαμε με τις προτάσεις αυτές λοιπόν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πρέπει να γνωμοδοτήσει με βάση τη συνθήκη και πολύ γρήγορα μετά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και, και την κατανόηση των κρατών μελών, του Συμβουλίου δηλαδή, που κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό του ε, δικαστηρίου και έπρεπε να πάρουμε ένα μέτρο ε, και το μέτρο αυτό ήταν η αύξηση ακριβώς του αριθμού των δικαστών. Ε, η πρόταση αυτή όμως δεν πέρασε προς το παρόν. Γιατί, Γιατί τα κρατημέλη, οι κυβερνήσεις δεν συμφώνησαν για τον τρόπο κατανομής των εδρών αυτών δικαστών. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως στο δικαστήριο, ε, το κοινοβούλιο μάλλον ε, μίλησε για, να, για την ύπαρξη καλών δικαστών. Τέλο πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι δεν υπάρχει και απόφαση από το 2011 μέχρι σήμερα. Τι συνέβη από τότε, το 2011. Καταρχά, ο αριθμό των υποθέσεων, των διαφορών που έχουν φτάσει ενώπιον του δικαστηρίου αυξήθηκε ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι αυξάνονταν στο παρελθόν. Σα είπαμε, στην περίοδο 2007-2013 ο αριθμό των υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου είχε αυξηθεί κατά 30% αυτό ο ρυθμός επιταχύνεται και επιταχύνθηκε και φέτος. Και για πρώτη φορά φέτος, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε πάνω από χίλιες υποθέσεις στις οποίες πρέπει να εγγύψουμε. Φυσικά το δικαστήριο εξακολουθεί να κάνει προσπάθειες για παραγωγικότητα. Προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, αλλά το δικαστήριο δεν καταφέρνει να ρυθμίσει, να διεκπαιρεώσει όλες αυτές οι υποθέσεις, όλο αυτόν τον όγκο υποθέσεων που λαμβάνει. Και επομένω, οι, οι υποθέσει υποθέσεις όλο και αυξάνονται. Υπήρχαν 3.300 εκκρεμεί υποθέσεις τη στιγμή που έκανε την πρόταση στο δικαστήριο και φέτος θα έχουμε 1.600 στο τέλος εκκρεμεί υποθέσεις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι δυστυχώ. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην, στο το δικαστήριο των Αμερικανών, ε, της Αμερικής, των ΗΠΑ, εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιες υποθέσεις είναι ε, σοβαρές και ποιες δεν είναι σοβαρές. Πρέπει να τις διεκπαιρεώσουμε όλες. Επομένως, ο σημαντικός αριθμός, η αύξηση του αριθμού των υποθέσεων ε, βαραίνει στο δικαστήριο και στην ε, λειτουργία του. Επίσης μιλούσαμε για τη διάρκεια των διαδικασιών. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Φυσικά η διάρκεια ε, δεν μπορεί να μειωθεί έτσι εύκολα λόγω του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που φτάνουν. Ε, υπάρχει και το οικονομικό θέμα, γιατί ξέρετε το δικαστήριο είναι υπεύθυνο για όλες τις οικονομικές διαφορές. Ε, υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, ε, κρατικών ισχύσεων, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, έχουμε δηλαδή υποθέσεις σε όλα αυτά τα επίπεδα. Αλλά για τις οικονομικές διαφορές ε, ανα ανταγωνισμό και κρατικέ ενισχύσει χρειαζόμαστε 48 μήνε. Τρία χρόνια δηλαδή. Πολύ χρόνο. Ακόμα χειρότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε πολλέ φορέ ότι η διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου ε, παραβιάζουν το άρθρο 47 της χάρτας λόγω της α, ε, παράλογης ε, διάρκειας των διαδικασιών. Και ενώπιον του δικαστηρίου αυτή τη στιγμή έχουμε προσφυγές οι οποίες εισήχθησαν γιατί θα πρέπει να... και ζητούν αποζημίωση διάφορες ας πούμε επιχειρήσεις λόγω της ε, πολύ μεγάλης διάρκειας της αρχικής δίκης. Το δικαστήριο ε, θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και θα απευθυνθεί τις επόμενες μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν, για να εξηγήσει την κατάσταση. Την κατάσταση που σας παρουσίασα συνοπτικά. Και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε μία λύση, ούτως ώστε να μπορέσουμε άμεσα να αποφασίσουμε άπαξ και διαπαντός α, ότι θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών που εκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου εδώ και 3,5 χρόνια. Το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως. Μπορεί να το επανεπιβεβαιώσει αυτό. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει αυτή την απόφαση. Και το δικαστήριο θα σα ανακοινώσει επίσης μια δεύτερη πρόταση νομοθετική, η οποία λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη, την οποία σας, παρουσίασα. Αυτή η δεύτερη νομοθετική πρόταση θα αποτελείται από δύο πτυχές. Από τη μία. Να φτάσουμε σε ένα διπλάσιο αριθμό δικαστών, δηλαδή στους 56. 56. Δηλαδή 28 συν 12 θα έχουμε 40 και θα προτείνει να προσθέσουμε ακόμη 16 ως 56, τόσο ώστε κάθε κρατός μέλος να έχει δύο δικαστές. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή της πρότασης. Δεύτερο στοιχείο, το δικαστήριο για τους δημόσιους υπαλλήλου θα πρέπει να εσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με αυτόν τον τρόπο θα έχει την απαραίτητη ισχύ για να ρυθμίζει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, όλες οι υποθέσεις που φτάνουν και, την... και τον αυξανόμενο ρυθμό ε, προσφυγών ενώπιον του δικαστηρίου και όλες τις διαφορές που υπάρχουν λοιπόν. Ε, όπως σας είπα, πρέπει να ληφθεί γρήγορη απόφαση για αυτή την πρόταση που υπάρχει εδώ και 3,5 χρόνια στο τραπέζι του νομοθέτη, του Συμβουλίου δηλαδή, και μια δεύτερη νομοθετική πρόταση που θα παρουσιαστεί με βάση το άρθρο 281 της ε, Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτή τη δεύτερη μεταρρύθμιση που θα συμπληρώσει το μηχανισμό ούτως ώστε άπαξ και διαπαντός το δικαστήριο να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που φτάνουν και που είναι κρεμείς, που, είναι, που έχουν φτάσει στο, στις πόρτες του και τις μελλοντικέ θα έχει την ε, δυνατότητα επίση το δικαστήριο σε λίγε εβδομάδε να σας παρουσιάσει σε μία συνεδρίαση με μία αντιπροσωπεία τη επιτροπή σα στο Λουξεμβούργο, εν πάση λεπτομερία όλα αυτά που θα διαβάσετε στα έγγραφα τα οποία θα λάβετε τι επόμενε ε, μέρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι για το δικαστήριο η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και ήγηκε η ώρα να ληφθεί μια απόφαση. Για το για να λειτουργεί απρόσκοπτα η δικαιοσύνη, για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών και για να λειτουργεί απρόσκοπτα η εσωτερική αγορά που είναι βασικό στοιχείο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, sir. Ευχαριστώ. Υπάρχει ο κύριος Φως που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά, έχω την αίσθηση ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση ερχόμαστε και αντιδρούμε με καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό. Έχουμε ένα σύστημα δικαίου, δικαιοσύνης, το οποίο λειτουργεί σωστά, είναι και η βάση για το κράτος ε, δικαίου που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει και να λειτουργεί σωστά. Και αν αφήσουμε αμφιβολίες ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και προβλήματα, τότε θα πληγεί και η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, διότι θα αναζητήσει κανείς άλλους δρόμους από το να περιμένει 4 ή 5 χρόνια για να εκδικαστεί μια υπόθεση. Οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντικό και από την άποψη του κράτους δικαίου, αυτό το στοιχείο δηλαδή που είναι το συνεκτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το καταστήσουμε και πιο λειτουργικό. Και όλα αυτά επηρεάζουν και την συνείδηση δικαίου που έχουμε. Πολλά κράτη-μέλη παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που αφορούν και τα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία όμως στη συνέχεια δεν ε, μεταφέρονται στις εθνικές νομοθεσίες σωστά. Όλα αυτά θα πρέπει να ε, μας επιστήσουν την ε, προσοχή στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί και ως προς τη δικαιοσύνη, ως προς το σύστημα δικαιοσύνης της. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα λειτουργικό σύστημα δικαιοσύνης και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε σε δύο επίπεδα μια λύση. Αφενός δηλαδή το δικαστήριο το ίδιο θα πρέπει να αναθεωρήσει και να ελέγξει τις δικές του διαδικασίες, πώς θα μπορέσει τις δικές του διαδικασίες με βάση και τις νομικές εγγυήσει και τις εγγυήσεις κράτους δικαίου για το πώς θα τις καταστήσει καλύτερες και στη συνέχεια θα μπορούσαν βεβαίως και να προσθεθούν και επιπλέον δικαστές. Τώρα αν θα είναι 12 ή 28, το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτήν την, ε, την ε, συσσόρευση υποθέσεων. Αν όμως τα κράτη-μέλη δεν μπορέσουν τα ίδια να ορίσουν τους, ε, τους δικαστές, τότε θα υπερβάλλω λίγο, ενδέχεται να δημιουργηθεί μια κατάσταση κατά την οποία ένα κράτος μέλος θα έχει πέντε δικαστές και ένα άλλο θα έχει μόνο έναν. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που πρέπει να ε, κρατήσουμε είναι ότι οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και κατά τη γνώμη μου όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ίδια, την, το ίδιο το σύστημα δικαιοσύνης που έχουμε και την ίδια τη συνείδηση περί δικαίου που δημιουργούμε στους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεπεδόν έχει το λόγο. Merci, le Ευχαριστώ. Εντάχει θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτό το αίτημα αύξησης του αριθμού των δικαστών κατά 12 ε, είναι υπερβολικό. Πρόκειται για πολύ μεγάλη αύξηση. Θα ήθελα να εξεύρουμε άλλα μέσα έτσι ώστε να εξοικονομήσει χρόνο το δικαστήριο. Στη Γαλλία εδώ και μερικά χρόνια είχαμε ένα παρόμοιο ε, πρόβλημα και βρήκαμε ένα φάσμα λύσεων για την επιτάχυνση της έκδοσης αποφάσεων και δεν ε, σημαίνει ότι θα επιλεγούν πραγματικά με αξιοκρατικά κριτήρια. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να τηρήσουμε τη σωστή κατανομή των δικαστών που να εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά ε, δικαστικά δικαιοδοτικά συστήματα. Δεν θα ήθελα η Γαλλία να βρεθεί σε μειονεκτική θέση μετά από αυτή την καινοτομία. Ο κύριος Κάστερ. αυτή η εξασφάλιση του κράτους ε, δικαίου είναι πραγματικά ένα κεντρικό θεμέλιο της ε, Ευρώπης, όπως είπε και ο κύριος Φως. Βεβαίως, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει και ένα λειτουργικό δικαστήριο. Και αν οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες, βεβαίως ε, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί αυτή, αυτή η αίσθηση κράτους δικαίου. Από αυτή την άποψη, η επιτάχυνση των διαδικασία... Ε, το αν αυτή η επιτάχυνση θα ενισχύσει την αίσθηση περί δικαίου, δεν, μπορώ, δεν θα ήθελα να το κρίνω. Σε κάθε περίπτωση ε, ενδέχεται και να υπάρχει ο κίνδυνος να, γίν, να εκδικάζονται υποθέσεις υπερβολικά γρήγορα και αυτό δεν θα είναι προς όφελος του συστήματος δικαίου και της δικαιοσύνης. Ακούσαμε ότι στις ΙΠΑ το ανώτατο δικαστήριο έχει 11 δικαστές. Εμείς έχουμε ήδη πολύ περισσότερους. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη διαφορά. Μήπως μπορεί κάποιο να μου ε, εξηγήσει σε τι οφείλεται η διαφορά αυτή. Επίσης έχω το εξής ερώτημα. Η αύξηση του αριθμού των δικαστών είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελβό. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμμερίζομαι όσα προελέχθησαν για την ε, σημασία του κράτους δικαίου ε, γιατί πρέπει να έχουμε, να διαθέτουμε ένα δικαστικό σύστημα που να είναι πραγματικά λειτουργικό. Δεν ξέρω γιατί στις ΗΠΑ λειτουργεί το σύστημα με 11 δικαστές, ενώ εμείς ε, χρειαζόμαστε, εμείς δεν τα καταφέρνουμε με 28. Ίσως το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο δεν μπορεί να αρνηθεί υποθέσεις, είναι υποχρεωμένο να δέχεται όλες τις υποθέσεις. Νομίζω όσον αφορά την ε, επαναδιοργάνωση, την εσωτερική επαναδιοργάνωση του δικαστηρίου, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για την πληθώρα υποθέσεων. Νομίζω ότι το δικαστήριο έχει προβεί σε ε, ε, μία επαναδιοργάνωση και έφτασε σε ένα κορεσμό. Άρα είναι πραγματικά σε απόγνωση οι δικαστές γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν τάσουμε υπέρ της αύξησης του αριθμού δικαστών και από όσο γνωρίζω θα υπάρχει αξιοκρατία, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Δεν μπορούμε να έχουμε πάνω από δύο δικαστές ανά χώρα. Υπάρχει αυτή η διτή προϋπόθεση. Τώρα με εκπλήσει η νέα πρόταση ε, διπλασιασμού του αριθμού των δικαστών ε, εκ των προτέρων μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ε, λειτουργούμε με 28, πολλοί θεωρούν ότι ήδη είναι πολύ. μετά προβάλαμε το ΣΥΝ 12 και τώρα γίνεται λόγος για διπλασιασμό. Μα δεν είναι καλό αυτό το μήνυμα που αποστέλουμε. Όλοι είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά δεν μπορούμε με το να ε, δρούμε με αυτόν τον πρωτογονισμό, δηλαδή με βάση τη χώρα προέλευσης. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πιέσουμε το Συμβουλίο ώστε να αποφασίσει την αύξηση κατά 12. Γιατί αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Νομίζω ότι γελιοποιούμαστε. Ευχαριστώ. Κύριος Καβαντά. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγκρίνω την ουσία των όσων προελέχθησαν. Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Καταρχήν, ένας από τους λόγους ε, για τον οποίο η Ευρώπη είναι πολύ μακριά από τον πολίτη, ένας από τους λόγους, υπάρχουν και πολλοί άλλοι, είναι ότι το δικαιοδοτικό σύστημα είναι πολύ αργό, δηλαδή 4 με 5 χρόνια για την επίλυση μιας διαφοράς. Είναι σαν να μπαίνουμε στη μάχη μετά από τη μάχη. Έγινε λόγος για το Αμερικανικό Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίζει τι ε, θα δεχτεί και τι θα απορρίψει. Αυτό δεν αφορά το ΔΕΚ, άρα δεν μπορούμε να κοιτάμε αυτό το πρότυπο, να προσβλέπουμε σε αυτό το πρότυπο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αποφαίνεται, υποβάλλεται μία ε, προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή. Άρα θα πρέπει να μπορεί να αποφανθεί πολύ γρηγορότερα. Δεύτερον, δεν είμαι ικανοποιημένος, όπως είπε και η κυρία Ντελβό, με το να διαθέτει κάθε χώρα δύο δικαστές. Είναι σαν να κάνουμε ένα patchwork. Δηλαδή τότε να ζητάμε ε, να έχουμε και τον ίδιο αριθμό επιτρόπων. Δεν ε, μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ε, είναι σαν να υποβαθμίζουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Είτε θα έχουμε ένα καθολικό δικαιοδοτικό σύστημα στην Ευρώπη και ο κύριος Λεπρετών έχει δίκιο θα πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα ή αλλιώς κατακερματίζουμε σε μικρά κομματάκια τυριού ε, ένα δικαιοδοτικό τρόπο δράσης και αντιμετώπισης των υποθέσεων. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει στενοπός καιρός είναι να την επιλύσουμε. Ο κύριος Σουσπάσκιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε όσα ήδη ακούστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να χάσει αυτό για το οποίο είναι εξαιρετικά περήφανοι. Ο κύριος Καβαντά είπε μόλις ότι η δικαιοσύνη απονέμεται μετά τον πόλεμο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν δικαιώματα και μπορούν να τα ασκήσουν, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε υπόθεση θα μπορεί να εκδικάζεται και μόνο στη συνέχεια να ε, λαμβάνετε απόφαση, να εκδίδεται απόφαση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο του συστήματος δικαιοσύνης που έχουμε. Thank you very much, uh, Mr. Buddha. Ευχαριστώ, κύριε Μπουντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρέμβω και να σε σχέση με αυτούς που λένε ότι δεν χρειαζόμαστε έναν επιπρόσθετο αριθμό δικαστών. Οι περισσότεροι είμαστε νομομαθείς και γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Πολλές φορές όμως εάν αποφαίνεται το δικαστήριο αργά δεν έχει νόημα. Τι θα κάνουμε όταν μας λέει το δικαστήριο ότι δεν τα καταφέρνει πλέον, θα το αφήσουμε να θαυτεί ή θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύσεις. Μία από τις λύσεις είναι η αύξηση του αριθμού των ε, δικαστών. Όσον αφορά τη, τα προσόντα αυτών των ανθρώπων, δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τα κράτη-μέλη δεν διαθέτουν δικαστές πραγματικά αποτελεσματικούς. Όμως, πολλές φορές μιλάμε για επιταχυμένες διαδικασίες. Εδώ δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάθε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μπορεί το δικαστήριο να αποφαίνεται ε, ως προς ε, το παραδεκτό των προσφυγών. Δεν μπορούμε να πούμε όμως τους δικαστές βρείτε τα, πρέπει να βρούμε λύσεις εμείς για να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε την ε, λειτουργία του δικαστηρίου. Ο κύριος Καλό τι σκέφτεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να παρέμβω για να μιλήσω για το ανώτατο δικαστήριο τον είπα, γιατί πρόκειται για διαφορετικό τύπο δικαστηρίου. Οι δικαστές στη Ουάσιγκτον δεν έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες ε, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όπως είπα εκείνοι μπορούν να επιλέξουν τις υποθέσεις που θα εκδικάσουν, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί να το κάνει. Άρα υπάρχει απροσπέλαστη διαφορά. Δεν ήθελα να σας επεξηγήσω σε λεπτομέρειες την πρόταση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όλες τις ε, λεπτομέρειες θα τις διαβάσετε και θα τη συζητήσετε με τα μέλη του δικαστηρίου και θα δείτε για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η δεύτερη διαδικασία που προανακοίνωσε το δικαστήριο. Εάν μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών με βάση την ε, πρόταση του δικαστηρίου, αυτό δεν οφείλεται στις ε, ενδοκυβερνητικές συζητήσεις για το ποιος θα εκπροσωπήσει ποιον. Το δικαστήριο το 2014 βρίσκεται σε μία πολύ πιο δυσχερή θέση από το 2011 και τώρα καταλαβαίνουμε ότι αν δεν κάνουμε κάτι τα επόμενα τρία χρόνια θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Έτσι εξελίσσεται η, έτσι εξελίσσεται η κατάσταση και αυτό θα σας επεξηγηθεί. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να βρουν λύσεις Η κυβερνήσεις. Η κατάσταση απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα, όπως θα σας εξηγήσουμε και κατά την επίσκεψή σας. Yes. Uh, Ο κύριος Μαρίνιο Πίντου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για να ξαναβάλουμε το πρόβλημα στις διαστάσεις του. Εμείς έχουμε καθυστερήσεις στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μία υπόθεση διαρκεί τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα υπήρξε η πρόταση αύξησης του αριθμού των δικαστών. Ίσως να είναι η πιο δαπανηρή λύση, αλλά και η πιο εύκολη. Εγώ όταν μίλησα για το ανώτατο δικαστήριο των είπα, ε, το ανέφερα για να πω ότι ένας δικαστής ε, θα πρέπει να έχει το κατάλληλο προσωπικό που να τον περιστοιχίζει. Το προσωπικό αυτό επιτελεί την εργασία σύμφωνα με τις κατευθυντηρίες γραμμές του δικαστή. Δεν θα ασχοληθεί με κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας ο ίδιος ο, δικαστής. Ένας δικαστής πλαισιώνεται και αποφαίνεται ως προς τη διαφορά καθεαυτή. Άρα το να αυξήσουμε αδιάκριτα τον αριθμό των δικαστών ίσως να μην είναι η καλύτερη λύση και δεν είναι και η λιγότερο δαπανηρή μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις που να απαλείψουν ορισμένες φάσεις της διαδικασίας, γιατί δεν είναι αποτελεσματικές, έτσι ώστε να αποφαίνονται οι ε, δικαστές ταχύτερα. Γιατί ε, διαρκεί μια υπόθεση τέσσερις, τέσσερα χρόνια. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια νομικήστικη προσέγγιση μία προσέγγιση ε, καθαρά τυπική ως προς τη διαδικασία. Υπάρχουν ε, ζητήματα που μπορούν να ε, επιληθούν πολύ πιο εύκολα από έναν γραφιά. Δεν χρειάζεται να παρέμβει ένας δικαστής. Άρα πρωταρχική μας, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να προστατεύουμε τον πολίτη που μας έχει εκλέξει. Μία δικαιοσύνη που καθυστερεί πάβει να είναι δικαιοσύνη. Όμως μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι τα αίτια της καθυστέρησης και της βραδιπορίας γενικότερα. Αλλά δεν μπορούμε να διασπαθίζουμε το δημόσιο χρήμα, το χρήμα του φορολογούμενου. Άρα θα πρέπει να διαγνώσουμε το πρόβλημα για να δούμε ποια είναι, ποιες είναι οι ρίζες ε, του κακού. Εάν ε, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι με την αύξηση των δικαστών επιλύουμε το ζήτημα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, προκαταλήψεις, ούτε συμφέροντα που να προωθούνται. Θα δούμε στη συνέχεια. Αν πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστών, καλώς. Αν μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις που απαλήφουν φάσεις της διαδικασίας που δεν έχουν λόγο ύπαρξης για να ε, αποφαινόμαστε, να αποφαίνονται οι δικαστές πιο γρήγορα, ίσως αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός τρόπος. Χρειαζόμαστε μία δικαιοσύνη που να δρά τάχιστα και να μπορεί να αποφαίνεται έγκαιρα ως προς τις διαφορές των επιχειρήσεων, των φυσικών προσώπων και της κοινωνίας γενικότερα. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία ανοιχτή. Ας γίνουν συγκριτικές μελέτες, διότι το θέμα με το ανώτατο δικαστήριο τον είπα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιλέγουν. Βεβαίως επιλέγουν, αλλά το ζήτημα είναι επί πόσων υποθέσεων αποφαίνεται ένας ε, δικαστής ετησίως. Να δούμε δηλαδή την αναλογία. Μιλάμε για 25 υποθέσεις ε, αναδικαστή είναι μια σωστή αναλογία ή όχι. Να δούμε τι συμβαίνει με άλλα δικαστήρια στα κράτη-μέλη και ίσως μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι οι δικαστές δεν είναι αρκετά παραγωγικοί. Αυτό συμβαίνει και σε αρκετά κράτη-μέλη. Άρα θα πρέπει να αναλύσουμε το ζήτημα, διότι ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως για κάθε δικαστή ε, θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσο είναι λογικό. Πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα. Και αν βάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία στο ζύγι και κάνουμε μία στάθμιση, θα δούμε εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε τη δικαιοσύνη, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και όχι τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Θα επισκεφθούμε το δικαστήριο, θα αναλύσουμε τα προβλήματα, θα μιλήσουμε με τους δικαστές και με το προσωπικό και θα βρούμε την καλύτερη λύση. Ο καθένας μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει, το δικαστήριο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λύσεις ε, για τις οποίες έχουμε προδικάσει την έκβαση. Ας γίνει σωστή διάγνωση και θα βρούμε την καλύτερη λύση για τους φορολογούμενους. Ευχαριστώ. Ε, thank you ε, Ευχαριστώ. Τελειώσαμε το σημείο αυτά λοιπόν. Και πάμε στο 9. Ο κύριος Σβιεύσκα έχει το λόγο. Πάρα πολύ έντονη και συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η συζήτηση για το πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η συζήτηση όλα, όλες αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να εξυπηρετούν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καλύτερη λειτουργία και από πλευράς δικαιοσύνης και από πλευράς οικονομικών, ούτω ώστε να έχουν ε, εμπιστοσύνη οι πολίτες στην ένωμη τάξη. Τώρα, για, το, για αυτό που θέλω να σας μιλήσω. Ε, το έγγραφο αυτό αφορά τον ίδιο στόχο, εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο. Μιλάει για τον κανονισμό για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας που εισήχθησαν το 2002 σχεδόν σε όλο το έδαφος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από μία χώρα, τη Δανία. Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται το αρμόδιο δικαστήριο και οργανώνει και την αναγνώριση των αποφάσεων αφαιρεγγιότητας. Μιλάμε φυσικά για τη διασυνοριακή αφαιρεγγιότητα εδώ. Το βασικό κριτήριο στη διαδικασία φερεγγιότητας που είναι και στοιχείο κλειδί, είναι το εξή. Αποφασίζουμε με βάση το ποιο είναι το κέντρο των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρεία για το ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο. Μέχρι στιγμής, ο ορισμός της βασικής έδρας της επιχείρησης ε, παραμελήθηκε λιγάκι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λιγάκι με τον ορισμό αυτό στο μέλλον, γιατί θα μπορούσε να μα βοηθήσει να επιλύσουμε κάποια προβλήματα. Στην πράξη τώρα, η βασική έδρα, η εταιρική έδρα, που αν θέλετε, είναι η βασική έννοια η οποία ανοίγει την πόρτα σε πάρα πολλές ερμηνείες, σε διαφορετικές συμπεριφορές, που μερικές φορές γύρουν προβλήματα. Ειδικά όταν μιλάμε για το λεγόμενο τουρισμό αφαιρεγγιότητας. Έτσι. Αυτή την ένθεση την εξηγήσω λίγο αργότερα. Θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με αυτό το κανονισμό περί αφαιρεγγιότητας. Η οικονομική κρίση, κυρίες και κύριοι, μας έπληξε τόσο, με τόσο τριμή τρόπο, ε, αισθανόμαστε ακόμη τις επιπτώσεις, που θεωρούμε ότι κάποια στοιχεία αυτού του κανονισμού εξακολουθούν να μην λειτουργούν όπως πρέπει. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να προσαρμόσουμε αυτόν τον κανονισμό στην ε, σημερινή κατάσταση και να εισάγουμε κάποιες αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια καλή λειτουργία της αγοράς. Της ενιαίας αγοράς δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός στόχος είναι η αλλαγή όλου αυτού του συστήματος, ούτως ώστε να αποφύγουμε το λεγόμενο form shopping την επιλογή δηλαδή του πλέον ευνοϊκού δικαστηρίου ή της καλύτερης δικαιοδοσίας. Θα πρέπει να έχουμε και μια πιο αποτελεσματική διαδικασία για την αφαιρεγκαιότητα ομίλου επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου αφαιρεγκαιότητας. Όλα αυτά τα βήματα θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να έχουμε μια πιο γρήγορη και πιο εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και να έχουμε μια καλύτερη εποπτική εικόνα της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Λένε στο παρελθόν, που ήταν πρόεδρος της νομικής ε, επιτροπής, είχε υιοθετήσει μία έκθεση, είχε γράψει μάλλον μία έκθεση και υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια το περασμένο Φεβρουάριο. Ε, η έκθεση αυτή συνοψίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Παράλληλα, το Συμβούλιο προσπάθησε να διαμορφώσει τη δική του άποψη για τον κανονισμό αυτό και ασχολήθηκε με το θέμα και υιοθέτησε την ε, θέση του τον Ιούνιο. Η θέση του Συμβουλίου επικεντρώθηκε καταρχάς ε, στο διατακτικό του κειμένου. Σήμερα η θέση του Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη και την αιτιολογική σκέψη και τα παρατήματα. Πρέπει να σας πω ευθύ εξ αρχής ότι οι θέσεις μας ημών και του Συμβουλίου διαφέρουν. Γι' αυτό ακριβώ, επειδή ακριβώ δεν ταυτίζεται η θέση μα, ετοιμάζουμε τη δεύτερη ανάγνωση, η οποία θα ξεκινήσει όταν το Συμβούλιο θα έχει υιοθετήσει το δικό του έγγραφο, που θα γίνει αυτό κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο. Δηλαδή, όσον ούπο. Αφού Ανάλυσα συνοπτικά και τα δύο έγγραφα, φτάνω στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι η θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου διαφέρουν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συγκλίνουμε καθόλου. Μπορούμε να φανταστούμε ένα συμβασμό ανάμεσα στα δύο όργανα. Το πιο βασικό είναι ο στόχος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι είναι ο ίδιος σε θέσει εργασία. Και είναι εξή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για την διαδικασία αφαιρεγγιότητας στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής Ένωση, η οποία θα μας επιτρέψει από τη μία να καλύψουμε τις ανάγκες των πιστωτών, πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε δηλαδή τα συμφέροντα των πιστωτών και παράλληλα, δεύτερον, έτσι, να μας επιτρέψει να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις που δυσκολεύονται, που είναι σε δυσκολία και που ενεργούν όμως τίμια. Προτείνουμε για αυτές τις επιχειρήσεις ένα σχέδιο, ε, ένα χρονοδιάγραμμα ε, μείωσης των, ε, χρεών, των δαπανών, των υποχρεώσεων δηλαδή, χωρίς να οδηγήσει όμως σε διάλυση της επιχείρησης, αλλά σε εξυγίανση της επιχείρησης για να προστατευτούν και οι θέσει απασχόληση. Είναι δικό μα στόχο και στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτό θα πρέπει να είναι βασικό στόχο κατά την αναζήτηση τη κοινή θέση σε δεύτερη ανάγνωση. Στο έγγραφο του Συμβουλίου υπάρχουν κάποιε νέε λύσει που δεν υπήρχαν στην πρόταση του Κοινοβουλίου. Είναι λύσει που αφορούν την χρεοκοπία ομίλου επιχειρήσεων, Και επίσης υπάρχει και η πρόταση για μια δευτερεύουσα διαδικασία και η πρόταση για μια συντονισμένη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις, μάλλον τις τρεις περιπτώσεις που σας απαρίθμησα, έχουμε τρεις εισάριθμες προτάσεις, τις οποίες πρέπει να εγγύψουμε, γιατί είναι προτάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του κανονισμού αυτού. Ένα στοιχείο κλειδί θα είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου που θα μας επιτρέπει ε, τη γρήγορη παρακολούθηση, γρήγορη ενημέρωση για τις διαδικασίες ε, αφαιρεγγιότητας που εκκρεμούν και είναι να εξελίξει σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να φτάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες και να μην υπηρετεί μόνο κάποιες αφηρημένες νομικές αξίες και έννοιες. Επίσης θα πρέπει να, να καταπολεμήσουμε τον τουρισμό αφαιρεγκαιότητα, όπως σας είπα. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του κανονισμού και την καλή επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου, ούτω ώστε όπως σας είπα να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πιστωτών. Νομίζω ότι οι λύσει που έχουν υιοθετηθεί προς το παρόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τι οποίε το... η βασική εταιρική έδρα είναι ο τόπος όπου ο πιστωτής έχει την οικονομική δραστηριότητα και είναι μια έξυπνη, ένας έξυπνος ορισμός και συνετός λογισμός, δεν υπάρχει λόγος να τον αλλάξουμε. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά την αφαιρεγγιότητα φυσικών προσώπων, την αφαιρεγγιότητα καταναλωτών δηλαδή. Είναι επίσης ένας τομέας όπου υπάρχει τεράστιο περιθώριο καταχρήσεων στα πλαίσια αυτού του τουρισμού αφαιρεγκαιότητας Και σε αυτή την περίπτωση η θέση μας με το Συμβουλίου είναι πολύ κοντά. Μια αποτελεσματική λύση σε αυτό το πρόβλημα διασυνοριακής αφαιρεγκαιότητας είναι απαραίτητη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση του τουρισμού και πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, θα μπορέσουμε να, να καταλήξουμε σε ένα κείμενο χρήσιμο με λίγη καλή θέληση από τις δύο πλευρές, γιατί εντάξει, χρειάζεται μια προσπάθεια για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Επίσης, κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει καλή θέληση, αλλά και το Συμβούλιο φυσικά, έτσι, προφανώς. Και ελπίζω από καρδιάς να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να φτιάξουμε ένα έγγραφο αποδεκτό και από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο και το οποίο θα είναι έτοιμο, ελπίζω, φέτος, μέσα στο 2014. Είναι απόλυτα ρεαλιστικό αυτό που λέω. Κύριε Πρόεδρε, να σα ενημερώσω ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελείται από τα εξή άτομα. Εγώ, εισηγητής, ο κύριος Κοφεράτη, ο οποίος θα εκπροσωπεί την ομάδα των σοσιαλιστών. Ο κύριος Ντούντα που θα εκπροσωπήσει τους συντηρητικούς. Ο κύριος Μάριο Πίντο από τους φιλελεύθερους. Η κυρία Καουτέλα, τους πράσινους. Δεν έχουμε ακόμα ε, πληροφόρηση για τον εκπρόσωπο της ομάδας EFD, δηλαδή της Ευρώπης της ε, ελευθερίας και της δημοκρατίας, ούτε πληροφορίες για το τι θα γίνει με την αριστερά, ποιος θα εκπροσωπήσει την ΚΟΕ. Ελπίζω να... Ευχαριστώ. Θέλει κανείς να βάλει το λόγο. Mr. Ράνιεφ. Κύριος Ράγγεφ. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Звиевка за подробно. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζιέφκα για την ε, λεπτομερή παρουσίαση του θέματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε χρόνο σχεδόν 200.000 επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρεοκοπούν και 1,7 εκατομμύρια άνεργοι προστίθενται στους ανέργους και δυστυχώς οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται. Γι' αυτό το λόγο θα χαιρέτιζα ε, μια γενική προσέγγιση του Συμβουλίου για τροπολογία του 1436 για τον εξυγχρονισμό της ε, διεκπαιρέωσης των ε, διαδικασιών αφαιρετικών σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις εθνικές διαδικασίες πριν από τις ε, διαδικασίες αφαιρεγγιότητας για να μπορούν οι επιχειρήσεις να ανακάμψουν και οι επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτά είναι θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το αν ε, η έδρα αυτεπάγγελτα μπορεί να ελεγχθεί ε, αυτό η, σε αυτό θα μια συντονισμένη διαδικασία αφαιροντικότητας θα μπορούσε να ε, οδηγήσει σε καλύτερη ε, ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για να διατηρούνται ε, καλύτερα οι ε, θέσεις απασχόλησης των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ και εγώ. Λέω Πρόεδρος, δεν υπάρχει κάποιος που έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Ζιεύκα θέλει να σχολιάσει. Ε, ε, Ωραία, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 10 και στο σημείο 11. Η συγγήτρια, η κυρία Βίξτρομ, ζητά συγγνώμη διότι προεδρεύει άλλης επιτροπής. Εκ μέρους της θα ανακοινώσω την ομάδα διαπραγμάτευσης που θα παρουσιαστεί ε, θα εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στους ε, τριμμές διαδρόμους. Είμαι εγώ από τους σοσιαλιστές, η κυρία Γκέριγκερ από το ΙΣΕΡ, είναι ο κύριος Ντούντα νομίζω, για τους φιλελεύθερους είναι η κυρία Βίξτρομ, από την ΚΟΕ είναι ο κύριος Μαξαλκάμ, από τους πράσινους ο κύριος Άντερστον, για το, την ομάδα EFDD είναι η κυρία Φεράρα. Η συγγήτρια προτείνει να γίνουν εσωτερικές συνεδριάσεις των σκιωδών συγγητών για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν τον επόμενο μήνα. Περισσότερες λεπτομέρειες ε, θα σας δοθούν σύντομα. Αυτά τα δύο, αυτά είχα να πω για τα σημεία 10 και 11 και μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 12. Το λόγο έχει ο κύριος Σάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην πραγματικότητα ε, μπορούμε να συζητήσουμε το 12, το 13 και το 14 μαζί. Είναι τρεις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για την ε, κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Υπάρχουν διάφορες, ε, διάφορα παράλληλα μέτρα από διάφορες παράλληλες διαδικασίες που θα ε, εξετάσουμε στο πλαίσιο αυτό. Τώρα έχουμε τρία ζητήματα και η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει αν αντιτίθεται το ένα φορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 το άλλο αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφορά 2, 3 και 8 και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 16, 24 και 38 και τα πρότυπα χρηματικής αναφοράς 3, 13 και ε, τα λογιστικά πρότυπα 40. Δουλειά της Επιτροπής μας τώρα είναι να αποφασίσει αν θα φέρουμε αντιρρήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι το Φεβρουάριο είχαμε υιοθετήσει τη δική μας θέση για, αυτή, για αυτές τις ε, προτάσεις όμνιμπους όπως αποκαλούνται της ε, Κομισιόν. Ωστόσο οι εργασίες ε, έχουν διακοπεί, υπάρχει αντίσταση στο Συμβούλιο. Δεν συνεχίζονται λοιπόν οι εργασίες, οπότε η Επιτροπή αποφάσισε να φέρει κάποιες τροποποιήσεις στη βάση της παλιάς διαδικασίας. Οπότε για αυτά τα τρία ζητήματα, για να μην ε, μπλοκαριστούν από το μεγάλο πακέτο, θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Άρα γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την παλιά διαδικασία και να κάνω μια γενική παρατήρηση, ότι είναι πραγματικά πολύ κρίμα που σταμάτησαν οι διαδικασίες η συνθήκη της Λισαβόνας ισχύει εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια και ακόμη δεν έχει ε, ευθυγραμμιστεί με αυτήν η διαδικασία που ακολουθείται, διότι το Συμβούλιο δεν θέλει να ε, παραιτηθεί των δικαιωμάτων του. Οπότε σε, σε τρεις μήνες ε, πρέπει να ε, υποβάλουμε την άποψή μας διότι τώρα έχουμε να κάνουμε με εκτελεστικές πράξεις αν μέσα σε τρεις μήνες ε, το Κοινοβούλιο δεν, ε, ή το Συμβούλιο δεν εκφράσουν αντιρρήσεις, τότε η Κομισιόν θα ε, εκδώσει αυτές τις εκτελεστικές πράξεις. Πρόκειται για μια πολύ ουσιώδη διαδικασία. Και η δική μου πρόταση είναι και για τα, και για τα τρία μέτρα να μην αντιτεθούμε να επιτρέψουμε δηλαδή στην ε, Κομισιόν να εκδώσει τις εκτελεστικές αυτές πράξεις. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ε, αντίρρηση ούτε από την πλευρά του Συμβουλίου, αλλά βεβαίως μπορούμε να χαράξουμε και μια δική μας ανεξάρτητη πορεία. Οι προτινόμενες ε, τροπολογίες αφορούσαν το, το περιεχόμενο δεν ε, ε, αντιτίθενται στην αρχή της ε, αυθεντικής ε, άποψης όπως είπε και η τεχνική γνώμη αφορούν τα, τα, τα κριτήρια της συγκρισιμότητας, της σταθερότητας που είναι τα, οι βασικές απαιτήσει, οπότε δεν υπάρχει ε, λόγος να αντιτεθούμε στην έκδοση και στην υιοθέτηση αυτών των ε, τροπολογιών. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που εμείς ε, προτείνω ως Επιτροπή να προχωρήσουμε την διαδικασία. Εντάξει, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο? Αν κατάλαβα σωστά, πρώτα απ' όλα προτείνεται να ψηφίσουμε από κοινού για τα τρία ζητήματα και μάλιστα μας καλύτερα να υπερψηφίσουμε. Αυτό που προτείνω είναι να μην αντιτεθούμε στα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν και για τα τρία θέματα αυτά. Ναι, αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο. Υπάρχει κάποιος που έχει αντιρρήσεις. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να ψηφίσουμε με ανάταση της χειρός και για τα τρία αυτά θέματα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχή. Ευχαριστώ πολύ. And we may go to point number. Και να προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 20 για την επικουρικότητα. Τον λόγο έχει η κυρία Δελβό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για κανονισμό του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εισαγγελικού Σώματος. Δεν είναι και πολυτεχνικό, έτσι, αλλά είναι πολύ πολιτικό. Πού βρέθηκε αυτό, καινούριο. Η υπεύθυνη κοινοβουλευτική επιτροπή για το θέμα είναι η Επιτροπή Δημοσίων και Πολιτικών Ελευθεριών. Μας αφορά ε, το θέμα γιατί 14, 14 κοινοβούλια από 11 κράτη-μέλη ε, απίφθηναν ε, μία αιτιολογημένη γνώμη ε, για το θέμα της επικουρικότητας. Η Κομισιόν απάντησε σε όλα τα επιχειρήματα αυτών των 14 εθνικών κοινοβουλίων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε νόημα να τροποποιήσουμε οτιδήποτε, γιατί η επικουρικότητα δεν υπησέρχεται. Το Κοινοβούλιο ε, ψήφισε ε, μια προσωρινή συμφωνία και ένα ψήφισμα. Είμαστε σε μια, στα πλαίσια μια ειδική νομοθετική διαδικασία. Υπάρχει αν υπάρχει συνένεση, μισό το να πρώτο άρθρο, με βάση το οποίο λειτουργούμε εν προκειμένου. Δεν το βρίσκω όμω. Είναι το άρθρο 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρχει συνένεση, στο εσωτερικό του Συμβουλίου το Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί. Αλλά δεν μπορεί να τροποποιήσει τίποτα, μπορεί να πει ναι ή όχι. Αν δεν υπάρχει συνένεση στο Συμβούλιο, τότε υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια ενισχυμένη συνεργασία. Χρειάζονται 9 κράτη-μέλη τα οποία θα συμμετάσχουν. Είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας, λοιπόν. Και επομένως κάποιες χώρες ε, είπαν εκ των προτέρων δεν, ότι δεν θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ το βρίσκω πολύ παράδοξο να πούν ότι δεν συμμετέχουμε, αλλά θα υποφεληθούμε παρόλα αυτά από τη διαδικασία της ε, κίτρινης κάρτας. για να βουλιάξουμε τον κανονισμό μέσω της επικουρικότητας. Προτείνω λοιπόν στην Επιτροπή δεν μπορώ να σας πω τη σωστή διατύπωση τώρα, αλλά να μην δεχτούμε αυτές τις αντιρρήσεις. Αυτό προτείνω ουσιαστικά. Να τους πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο, ότι δεν μπορούν να παρέμβουν. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στα χέρια της ε, Κομισιόν τώρα. Μια και η Κομισιόν απάντησε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας ε, πρόκειται να λάβει υπόψη τι γνωμοδοτήσεις των κρατών μελών, τις απόψεις των κρατών μελών και το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ζήτησε να γίνουν ε, συστάσεις προς την Κομισιόν με κάποιες διευκρινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην πραγματικότητα είναι κάτι θετικό. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη, έτσι. Αυτό θα υλοποιήσει, αυτό θα κάνει η εισαγγελία. Δηλαδή μπορεί να διώξει σε περίπτωση που ε, υπάρχει ζημία απέναντι στα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμω να έχουμε το μέρο μα και του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω λοιπόν από την Κομισιόν να μην κάνει τίποτα και να περιμένουμε τη συνέχεια τη διαδικασία. Δηλαδή να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Πολύ απλά. Θέλει κανένα το λόγο. Δεν νομίζω. Ήταν το τελευταίο σημείο αυτό στην πρωινή μας συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα με το εργαστήρι μας και αύριο θα αρχίσουμε στις 10.30 το πρωί γιατί έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών σήμερα. Έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα μέχρι τις 11.30 και εν συνεχεία θα συνεχίσουν οι συντονιστές στη συνεδρίασή τους. Σας ευχαριστώ. May Όσοι δεν έχουν δουλειά εδώ, παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα γιατί η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα και κλεισμένο των θυρών.